Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, σα παρακαλώ, καθίστε στι θέσει σα. Συνεχίζει τη συνεδρίαση. Έχω τα αποτελέσματα των εκλογών. Εκλέγοντες. 713. Ε, Λευκά ή άκυρα

Συγχαρητήρια κύριε Μπούσεκ Λίβε Αγαπητοί συνάδελφοι. Συγχαρητήρια κύριε Μπούζεκ, λέει ο πρόεδρος στα ε, πολωνικά. Σας συγχαίρω για την επιτυχία σας. Πρώτα είμαι πολύ σημαντική θέση και σας συγχαίρω για την επιτυχία σας αυτή. Κυρία Εύα Μπριτ Σβένσον πήρε 89 ψήφους. Άρα ο Γιώργη Πουτσέκ ε, πέτυχε την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων. Και αυτό που είπα στα πολωνικά, προσπάθησα να πω μόλι τώρα στα πολωνικά, θα σα το πω και στη δική μου γλώσσα συγχαίρω εγκαρδιότατα το Γερσί Μπούσεκ για την ε, εκλογή του που είναι τόσο πιστική. Του εύχομαι κάθε επιτυχία για το θαυμάσιο αυτό έργο που αναλαμβάνει τώρα. Και τον παρακαλώ να έρθει εδώ στο θόκο του Πρόεδρου. Παρακαλώ, αγαπητέ Γερσί Μπούσεκ. Koleżanki i koledzy, dear colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας ευχαριστήσω που με εξελέξατε πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι και μια τεράστια τιμή, αλλά και μια πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα αυτή η εκλογή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι με υπερψήφισαν. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μην σας απογοητεύσω και για αυτούς οι οποίοι δεν ψήφισαν το άτομό μου θα προσπαθήσω να σας πείσω ότι θα εργαστώ με όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου ανεξάρτητα από την πολιτική παράταξη στην οποία ανήκουν και βασίζομαι στην υποστήριξή σας. Ευχαριστώ και την κυρία Σφένσον, η οποία έλαβε μέρος στις εκλογές του Προέδρου και για όλες τις συζητήσεις που είχαμε μαζί. Για όλους τους συναδέλφους μας και ιδίως στον αναφερόμενο στον Μάριο Μάουρο και τον Γκρά